Ladies and gentlemen, uh, good morning. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, σας παρακαλώ καθίστε, αρχίζουμε αμέσως την συνεδρίαση, δηλαδή την το δεύτερο μέρος ε, της συνεδρίας αυτής με την έγκριση της ε, ημερησίας διατάξεως να έχει γίνει ήδη από χθε και τώρα είναι το θέμα ο αγώνας κατά της πειρατείας Τη θάλασσα γύρω από την Αφρική. Έχω τρει πάνελις, τον κύριο Βαντερ Α, ακόμη δεν έχει φτάσει, όμω αν του έρχεται. Καθίστε παρακαλώ. Θα ήθελα να απευθύνω το καλώς ορίσατε στους τρεις πανελίστ. Πρώτος είναι ο κύριος Άλαν Κόουλ, της UNDAC από το Περιφερειακό Γραφείο του Διεθνούς Προγράμματος Αντιμετώπισης του Εγκλήματος με ειδικότητα στην Ανατολική Αφρική. Δεύτερος είναι ο κ. Μάρκους Χούμπεν που εκπροσωπεί την EEAS δηλαδή την ομάδα επαφών για την πειρατεία και ο, το τρίτο μέλος του πάνελ είναι ο κύριος Βάντερ Πέλ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Κόλ για να αναπτύξει το θέμα που έχουμε στην ημερήσια διάταξή μας. Έχετε το λόγο κύριε. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνετε να απευθύνουμε το λόγο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το έργο που κάνει το Γραφείο Εγκλήματος και Ναρκωτικών των Ηνωμένων Εθνών που έχει αρχίσει να εμπλέκεται στον αγώνα κατά της πειρατείας αρχικά μόνο για την Σομαλία από το 2009. Αυτή η εμπλοκή μας χαρακτηρίζεται από πολύ στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα μέρη της. Το γραφείο μας των Ενωμένων Εθνών είναι τμήμα της Γενικής Γραμματείας των Ενωμένων Εθνών. Είμαστε εξειδικευμένος οργανισμός με εντολή να αντιμετωπίζουμε κατά πολέμηση ναρκωτικών, ε, οργανωμένου εγκλήματος και πειρατείας. Εμένα ειδικά με ενδιαφέρει το διεθνές έγκλημα στην θάλασσα. Ο καλύτερος τρόπος για να εξηγήσω πόσο έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και η συνεργασία μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να δώσω με λίγες γραμμές τα χαρακτηριστικά της δουλειάς μας και στην Ανατολική Αφρική. Πρώτα, επισημαίνω τη στενή μας διασύνδεση με τις ναυτικές δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια υψηλή απόδοση αποστολή στον ε, Ινδικό ωκεανό. Έχουμε συνεργαστεί πολύ στενά. Το έργο μας περιλαμβάνει και την ανάπτυξη κέντρων εκδίκασης των υποθέσεων σε χώρες όπως οι Σεϊχέλες για να διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν τόποι όπου μπορούμε να παραδώσουμε τους υπόπτους πειρατείας για να δικαστούν. Σε στενή διαβούλευση βέβαια με την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό ο μηχανισμός που λειτουργεί είναι ότι οι ναυτικές δυνάμεις της Ένωσης παραδίδουν τους υπόπτους πειρατείας σε τέσσερις τόπους όπου το, τα Ηνωμένα Έθνη ενισχύουν τις τοπικές αρχές για να ασφαλιστεί δίκαιη δίκη και βέβαια ανθρώπινες συνθήκες κράτησής τους. Το έργο αυτό, όπως είπα από το 2009, υποστηρίζεται από το Instrument for Stability και έχουμε υποφερθεί και εμείς από το όργανο αυτό στην Κένια, σε Ιχέλες και στον Μαυρίκιο. Να επισημάνω ότι η πρόκληση της διασφάλισης ότι ένας νεαρός ύποπτος πειρατείας μεταφέρεται σε, σε κράτος της περιφέρειας, όπου όμως ισχύουν όλες οι προδιαγραφές της δικαιοσύνη που ε, πρεσβεύουν τα Ηνωμένα Έθνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό αυτό. Χωρίς τη συνεργασία αυτή δεν θα ήταν δυνατό να προσφέρουμε σήμερα την εξασφάλιση στο Κοινοβούλιο σας ότι όλα τα πρόσωπα αυτά τα οποία μεταφέρονται και παραδίδονται εκεί αντιμετωπίζουν δίκη, δίκαιη και που να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Έχουμε και το προγραμμάσι στον Ειδικό Ωκεανό για την διασφάλιση ότι οι ίδιες χώρες που συνεργάζονται με το Γραφείο των Εθνών έχουν λειτουργικά συστήματα απονομής δικαιοσύνης που να εξασφαλίζουν ότι όχι μόνο η πειρατεία αλλά και άλλα ναυτικά αδικήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν. Στην ίδια τη Σομαλία συνεργαζόμαστε στενά με την οργάνωση με της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι κατεστημένη εκεί για εκπαίδευση προσωπικού και σε λιμάνια και βεβαίως και με τον απαραίτητο εξοπλισμό. Τέλος, θα ήθελα να μιλήσω και για την ομάδα επαφών για την πειρατεία που αποτελεί και πρότυπο διεθνούς συνεργασίας και με τον, τους ενδιαφερόμενους κλάδους αλλά και με τις αρμόδιες οργανώσεις. Και ο κύριος Χούμπεν θα αναπτύξει περισσότερα τα πράγματα αυτά. Από τη δική μας σκοπιά εμείς υποστηρίζουμε τη νομική εργασία που γίνεται εκεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ίσως θα ενδιαφερθεί να μάθει ότι διεξάγεται πολύ καινοτόμα νομική εργασία όπου περιλαμβάνονται και απαραίτητες ρυθμίσεις για την μεταφορά των Σομαλών υπόπτων πειρατείας από τα πολεμικά σκάφη στην ξηρά για πρόσωπα που είναι κάτω των 18 ετών απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη μεταχείριση η μεταφορά των κρατουμένων στην ίδια τη Σομαλία όπου προβλέπονται και ε, Υπάρχουν και εγκαταστάσεις μάλιστα για μακρόχρονη κράτησή τους, καθώς και το απαραίτητο προσωπικό. Τώρα για την Δυτική Αφρική. Εδώ περισσότερο το θέμα είναι ένοπλης ληστείας με πολλές ε, περιπτώσεις επιθέσεων. Εκεί είναι πιο στενό το έργο μας, είναι τα νομικά πλαίσια και η εκπαίδευση του προσωπικού δικαστικού αστυνομίας. Εκεί η Ιντερπολ και άλλοι εξετάζουν την επιβολή του νόμου στην ξηρά, καθώς και άλλες προκλήσεις. Στη Δυτική Αφρική αντιμετωπίζουμε εγκληματικά καθεστώτα, τα οποία δεν αντιμετωπίζουν αυτά τα αδικήματα. Χρειάζεται εξυγχρονισμό ο τρόπος αντιμετώπισης, χρειάζεται πολύ, πολύ καλύτερη επικοινωνία μεταξύ χωρών μελών και τοπικών περιφερειακών οργανισμών και εκεί κάνει πολύ σημαντική δουλειά η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών. Ως υποσημείωση αναφέρω και την Νοτιοανατολική Ασία, στην οποία έχουμε σημαντικό, σημαντικότερο αριθμό πειρατιών και από την Ανατολική Δυτική Αφρική. Πρόσφατα επιστρέψαμε από Ινδονησία και Ταϊλάνδη όπου συνεργαστήκαμε για να αναπτυχθεί εκεί ένα πρόγραμμα. Τα κέρδη είναι τεράστια από την πειρατεία στη Σομαλία και αυτά έχουν χαρίνει και άλλους σε άλλα μέρη του κόσμου να προσφύγουν σε αυτόν τον τρόπο πρόσκλησης κερδών. Σε ό,τι αφορά τώρα το μέλλον, έχω τις εξής ας πούμε προσεκτικές παρατηρήσεις να κάνω. Δεν θα πρέπει να υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η πειρατεία μπορεί να επανέλθει στην Ανατολική Αφρική. Έχουν περάσει δυόμιση χρόνια από την τελευταία επίθεση. Όμως οι συνθήκες που υπήρχαν το 2007 και 2008 όταν άρχισαν οι πειρατικέ επιθέσει, εξακολουθούν να υπάρχουν. Πολλοί νεαροί Σομαλοί που έχουν πρόσβαση σε όπλα και σε σκάφη, πολλά μεγάλα σκάφη περνούν κοντά από τι ακτέ τη Σομαλίας και επιχειρήσεις, ναυτο, ε, ναυτικές επιχειρήσεις οι οποίες είναι διατεθειμένες να πληρώσουν λίτρα για τα πλοία και για τα πληρώματά τους. Υπάρχουν λοιπόν όλες οι συνθήκες οι οποίες υπήρχαν ήδη το 2007 και το 2008, εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα. Τούτου λεχθέντος έχουμε δει βέβαια σημαντικότατη μείωση του αριθμού των πειρατιών και του τελευταίους περίπου 30 μήνες χάρη στην, στον επιτυχημένο συνδυασμό και των ναυτικών επιχειρήσεων και ε, της δράσης επιτόπου, βελτίωση και της διαχείρισης επί των πλοίων βλέπουμε από τις εκθέσεις του προσωπικού μας που είναι, έχει έδρα σε πέντε ε, μέρη της Σομαλίας ότι έχουν μειωθεί. Τώρα, τελευταία παρατήρηση τώρα για την Ανατολική Αφρική. Υπάρχουν 26 όμοιροι ακόμα στην Σομαλία από έναν αριθμό 750 κάποτε. Μόλις καταφέραμε να ε, συμβάλλουμε στην απελευθέρωση άλλων τεσσάρων που είχαν κρατηθεί εκεί μια πενταετία και βεβαίω πέρασαν απίστευτε δυσκολίε και στερήσει σε αυτά τα πέντε χρόνια. Εκτό από του 26 ομήρου που κρατούνται ακόμα στην Σομαλία, έχουμε 1.400 Σομαλού πειρατέ και υπόπτου που κρατούνται σε φυλακέ 21 χωρών σε όλο τον κόσμο. Ελπίζω ότι αυτά τα στατιστικά στοιχεία σα δίνουν και μια ιδέα της προσπάθειας που έχει κάνει το γραφείο μας των Εθνών αλλά και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο αριθμός των 21 χωρών ανα, ανα τον κόσμο όπου κρατούνται ε, είναι και αυτό μια σημαντική συνεργασία. Παρόλο που είδαμε μείωση της πειρατείας στην Ανατολική Αφρική και είπα προηγουμένως ότι μπορεί και να συνεχίσει να αυξάνεται ωστόσο στη Δυτική Αφρική και στην Ανατολική Ασία Παρ' όλα αυτά, οι θάλασσε του Ινδικού ωκεανού δεν έχουν απαλλαχθεί από εγκληματικέ ενέργειε. Στου τελευταίου έξι μήνε στην Ανατολική Αφρική βρέθηκε παραπάνω ηρωίνη στην θάλασσα από τα τελευταία 20 χρόνια. Στην Κένια βλέπουμε τώρα την ηρωίνη να καταναλώνεται περίπου σε ποσό 2,5 τόνων ε, ε, επιτοπίω και το δεκαπλάσιο διακινείται. Αυτό με εμπλοκή και όσων εμπλέκονται και στην πειρατεία, οι οποίοι τώρα ε, προχωρούν και στο λαθρεμπόριο ηρωίνης και όπλων και μεταναστών. Υπάρχουν δηλαδή εγκληματίες οι οποίοι θα δράξουν κάθε ευκαιρία που τους προσφέρεται. Το ίδιο στην Ανατολική Αφρική το 2010 είδαμε εκατομμύρια δολάρια να περνούν, αξία δηλαδή, ε, τέτοιο λαθρεμπόριο να περνά προς την Ευρώπη. Πολλά από τα εγκλήματα που συμβαίνουν εκεί τελικώς το τελικό τους αποτέλεσμα συμβαίνει στην Ευρώπη. Ελπίζω να σας έδωσα να κατανοήσετε το πού βρίσκεται η πειρατεία αυτή τη στιγμή στην Ανατολική Ασία και στην Δυτική Αφρική. Εξακολουθεί η στενή συνεργασία μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. είναι πολύ περισσότερο μια στενή εταιρική σχέση και συνεργασία μέσα στην τελευταία εξαιτία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε αυτά τα σχόλιά μου. Ευχαριστούμε κύριε Κούλ. Σίγουρα θα υπάρξει πολύ ε, περισσότερος χρόνος κατά τη συζήτηση. της To, to... Ώστε να δοθούν απαντήσει. σε ερωτήσει και παρατηρήσεις για αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Ο κύριος Κούμπεν τώρα, παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, κύριε και κύριοι, σα ευχαριστώ για την πρόσκληση σήμερα να μιλήσω για την πειρατεία στην Αφρική. Θα ήθελα να σας δώσω κάποιες ε, πληροφορίες ε, για την ε, οργάνωση και το συντονισμό της διεθνούς ανταπόκρισης απάντησης στα φαινόμενα αυτά. Ιδιαίτερα την CGPCS, δηλαδή την ομάδα, την ομάδα επαφής και συντονισμού, η οποία συνομαδοποιεί όλους τους ενδιαφερομένους ε, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ε, ε, πολιτικούς και στρατιωτικούς. Πρόκειται λοιπόν για μια δομή που αντιπροσωπεύει ένα νέο διακυβερνητικό διεθνές πρότυπο για νέες προσεγγίσεις σε περίπλοκα διεθνή προβλήματα. Η ομάδα επαφής λειτουργεί συνεχώς από το 2009 και ήταν Ουσιαστική σημασία για να επιτευχθούν κάποια απτά και συγκεκριμένα θετικά αποτελέσματα. Επί τη βάση του ότι, όπως είπε και ο πρώην πρόεδρος της ομάδας επαφής, κανείς ε, ε δεν συμπαθεί τους πειρατές. Υπάρχει μια ομοφωνία επ' Έχουμε λοιπόν μια ασυνήθιστα ανοιχτή αρχιεκτονική δομή με φορεί που είναι διατεθειμένοι να συνεισφέρουν σε λύσει για την υπηρετία, μεταξύ των οποίων ε, κυβερνητικού φορείς, ε, περιφερειακούς ε, μη κυβερνητικού φορείς, με εκπροσώπηση των ναυτιλιακού κλάδου, μια μοναδική δομή γιατί δεν υπάρχει επίσημη <clears throat> νομική δομή, πρωτόκολλο, μόνιμη δομή, δεν υπάρχει θεσμική ομπρέλα θέλετε. Δεν υπάρχει γραμματεία, δεν υπάρχουν επίσημοι κανόνες για μια μεταβατική δομή ε, πολιτικής ε, εθελοντικής συμμετοχής και έχει μια πολύ εστιασμένη και περιορισμένη ε, προσέγγιση για την πειρατεία <clears throat> στα, έξω από τα ύδατα της Σομαλίας. Με τη συνεργασία διαφόρων φορέων που κανονικά δεν θα συνεργάζονταν μεταξύ τους ε, σε τόσο υψηλό ενδιαφέρον. Η ομάδα επαφή συνεργάζεται με τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά δεν ανήκει, δεν υπάγεται στα Ηνωμένα Έθνη. Και αποδίδει. Υπήρξε σημαντική για να δώσει απαντήσεις στα φαινόμενα και να περιορίσει τα φαινόμενα της πειρατείας σχετικά με τη μεταφορά των υπόπτων για παράδειγμα προς τις Ιχέλες και εφόσον κατεδικαστούν τον επαναπατρισμό τους στη Σομαλία για την κράτησή τους. Επίση ε, διοργανώθηκαν εθελοντικές ε, επιχειρήσεις θαλάσσιες ε, των λεγόμενων independent deployers. Η ομάδα επαφής επίσης έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο για ενδιαφέρουσα συνεργασία με τον κλάδο της αφιλίας προκειμένου να διευκολύνει την δίωξη των διοργανωτών και των χρηματοδοτών των εγκληματικών αυτών οργανώσεων Επίσης ε, υπήρξε σημαντική σε μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης ε, ιδιαίτερα για τους νέους της να αποφεύγουν τη συμμετοχή τους σε τέτοιες ομάδες. Είναι λοιπόν ε, σωστό να πει κανείς ότι έχει πετύχει μια πολιτική νομιμοποίηση η ομάδα επαφή χωρί να, έχει ομάδα, χωρίς να έχει επίσημη δομή, όπω σα έλεγα, γιατί βασίζεται στην εμπιστοσύνη. Η συνεργασία αυτή <clears throat> επί μακρό χρονικό διάστημα έχει οδηγήσει σε συνέργειες και κοινή κατανόηση και ιδιαίτερα το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών, το UNODC, ήταν πολύτιμο συνεργάτη. Θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω και να χαιρετήσω τον κύριο Άλαν Κόουλ που προσωπικά ενέχεται και είναι πρότυπο τη έξοχη αυτή συνεργασία που έχουμε στα ύδατα τη Ευρική για την καταπολέμηση πειρατεία. Τώρα να σα πω ε, δύο λόγια για την Προεδρία τη Ευρωπαϊκή Ένωση τη Ομάδα Επαφή. Η Ένωση ήταν παρούσα από την αρχή από τότε κάναμε μια ε, εντυπωσιακή πορεία. Αρχικά ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν παρατηρητής. Ε, τέσσερα χρόνια αργότερα προσεκλήθη να αναλάβει την Προεδρία από τον Ιανουάριο του 2014. Ο κύριος Μάτσικ Ποπόσκι, ε, Γενικός Γραμματέας της υπηρεσίας that e της e θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω επίσης ότι η ΓΔ Move και ΔΕΦΚΟ ιδιαίτερα ο πλευράς της Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Εκπροσώπηση στη Νέα Υόρκη, η UNAF στην Αταλάντα, αν ακούσαμε καλά τον ομιλητή, εν πάση περιπτώσει, ε, επί τη αρχή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν <clears throat> εκπροσωπείται ενιαία και όχι από τους ε, μεμονωμένους ε, θεσμούς ή οργανισμούς της. Όλοι αυτοί συνεργάστηκαν προκειμένου να γίνει η, ομάδα επαφή επιτυχής. Είχε θέσει ένα φιλόδοξο στόχο μάλιστα. Ο πρώτος εκ των οποίων είχε αποτυπωθεί ω 0-0. <clears throat> μηδέν επεισόδια και μηδέν σκάφη στα χέρια των πειρατών. Επίσης η ομάδα επαφής έπρεπε να γίνει πιο αποτελεσματική ως προς το κόστος και να ε, εστιάζεται στην ζήτηση, δηλαδή στην ανάγκη επίλυσης συγκεκριμένων προβλημάτων. Επίσης έχουμε ε, προετοιμάσει ένα έγγραφο με πορίσματα του τι και πώς κάναμε και πώς λειτουργήσε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε μηδέν σκάφη στα χέρια των πειρατών από τα 60 που είχαμε το 11 η ναυτική εχμάλωτη από 750 έχει κατέλθει ο αριθμός τους σε 26 μόλις το Μάρτιο του 2015. Οι τελευταίοι απελευθερώθηκαν πριν από ένα μήνα μετά από τεράστια και δυσάρεστη προσωπική περιπέτεια. Ο Γενικός Γραμματέας χαιρέτησε το κουράγιο τους και ζήτησε την άμεση απελευθέρωση των 26 υπολείπων ομήρων. Τον Οκτώβριο του 2014 η ομάδα επαφής συνέστησε μια Piracy Survival Family Fund, ένα ταμείο κοινωνικής υποστήριξης και προστασίας των οικογενειών των ναυτικών αυτών, των θαλασσοπορών που είναι εκμάλωτοι. Επανερχόμενος τώρα στη δομή, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήθελε να, γίνει, να εστιάζεται στις ανάγκες. Ε, τα μέλη έχουν τι από 5 σε 3 και το νομικό φόρουμ ε, με συμπροεδρία Πορτογαλίας και Μαυρικίου επιτρέποντας λοιπόν τις χώρες της περιοχής της ευρύτερης να αναλάβουν την ευθύνη όχι μόνο των προβλημάτων και της επίλυσής τους με ενεργή ρόλο της ε, Επιτροπής του Ινδικού Κόλπου, των, ε, της ομάδας επαφής των Αραβικών ε, Εμμυράτων μεταξύ άλλων. <clears throat> Επίσης έχουμε εστιαστεί στα, στις εμπειρίες που έχουμε συσσωρεύσει από αυτή την προσπάθεια προκειμένου να ενημερώσουμε τους πολιτικούς ηθήνοντες και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Ένα κονσόρτιουμ επίσης συνεστήθη από ερευνητές ε, του Πανεπιστημίου του Κάρντιφ και έχει ολοκληρωθεί ένα πρώτο στάδιο ανάλυσης επί της ομάδας επαφής. Θα ήθελα ιδιαίτερα να αναφερθώ στα μέλη της Επιτροπής μια δημοσίευση υπό το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο ε, Μελετών Ασφαλείας ε, το Genesis αν ακούσαμε καλά. Επίσης ε, κάποια σχόλια για ένα ακαθόδες ζήτημα, δηλαδή την επανεξέταση της ε, λεγόμενης περιοχής high risk ε, στον Ινδικό ωκεανό. Έχουμε μια ομάδα χωρών μεταξύ των οποίων Αίγυπτος, Πακιστάν, Σαουδική Αραβία, Ομάν, Τζιμπουτί, που ζητούν επανεξέταση, αναθεώρηση της περιοχής αυτής του ψηλού Από την άλλη, ο ιδιωτικός τομέας της ναυτιλίας θέλει να διατηρήσει την, αυτή την περιοχή όπως ε, υψηλού κινδύνου που περιγράφεται αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται λοιπόν να καθορίσουμε ένα κοινό τρόπο προς τα εμπρός, μια κοινή λύση. Είναι προφανές ότι η απόφαση της επανεξέτασης αναθεώρησης εξαρτάται πολύ από τον κλάδο, αλλά <clears throat> και μη και φορείς που δεν θα προέρχονται από τον κλάδο θα πρέπει να ενέχονται στην επανεξέταση αυτή. Ο κ. Ποπός και όπως με επικεφαλής της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ηγείται των προσπαθειών μεταξύ των οποίων συναντήσεων που έγιναν την περασμένη εβδομάδα ώστε να βρεθεί μια λύση στο ζήτημα αυτό στο άμεσο μέλλον. Κυρίε και κύριοι, στα τελευταία λεπτά έχω χαιρετήσει τις προσπάθειες της ομάδας επαφής ε, για την πειρατεία. Πρόκειται για ένα πρότυπο επί τη βάση της ανάλυσης του κινδύνου. Ε, θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Προεδρία ήταν σημαντική και σημαδιακή θα έλεγα, γιατί για πρώτη φορά διεθνής οργάνωση και όχι κυβέρνηση εθνική ε, έχει την Προεδρία. Επίσης είναι ένα πρότυπο ε, και ένα πλαίσιο επίλυσης προβλημάτων διεθνούς συνεργασίας. Η ομάδα επαφής έχει επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει διεθνή ευθύνη και να ηγηθεί στην προσπάθεια αυτή διευκολύνοντας το συντονισμό ε, μια ομάδα τελείω διαφορετικών φορέων ενδιαφερομένων προκειμένου να εξευρεθούν λύσει. Η ίδια η φύση τη Ευρωπαϊκή Ένωσης μας δείχνει πόσο σημαντική είναι η πολυμέρεια, είναι στο γενετικό μας κώδικα στην Ευρώπη. Τα 28 αυτά κράτη-μέλη που είναι η επιρροή του πολύ σημαντικότερη από την επιρροή που θα μπορούσε να έχει οποιαδήποτε χώρα από μόνη της. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο η ομαδοποίηση όλων αυτών των ενδιαφερομένων φορέων στην ομάδα επαφή είναι πολύ πιο ε, επιρροή επιρροής από αυτή που θα μπορούσαν να έχουν οι φορείς. Ε, σας ευχαριστώ. Τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Άντιαν Φάντερ Μέρ της ε, ΓΔ ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ε, αγαπητοί βουλευτέ και συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ενημερώσω για μία σειρά από δράσεις τις οποίες έχουμε εφαρμόσει και οι οποίες συνεχίζουν να εφαρμόζονται στο πλαίσιο της καταπολέμησης της πειρατείας ε, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Θα ήθελα καταρχήν να σας ε, υπενθυμίσω ότι το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2008, το οποίο υπήρξε πολύ σημαντικό, για όλους μας ως μια κατευθυντήρια γραμμή ε, προκειμένου να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας ε, προς αυτή την κατεύθυνση εξακολουθεί να παραμένει επίκαιρο ε, και σήμερα σε ό,τι αφορά την κατάσταση, σε ό,τι αφορά την πειρατεία και την ευαισθητοποίηση σε ό,τι αφορά την πειρατεία. Και θα ήθελα να αναγνωρίσω αυτές τις συνεισφορές γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι σήμερα να ξέρουμε ε, πού βρίσκονται τα πλοία και να εντοπίζουμε τις ε, κινήσεις οι οποίες μπορούν να μας ε, οδηγήσουν στο να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει κάποια δραστηριότητα από πλευράς πειρατική δηλαδή. Επίσης θα ήθελα να τονίσω εδώ ότι η πειρατεία αποτελεί τον τελευταίο κρίκο μιας ολόκληρης αλυσίδας. Δηλαδή πρόκειται για μια δραστηριότητα η οποία σχετίζεται με το οργανωμένο έγκλημα, κάτι το οποίο θέλουμε να προλάβουμε εφαρμόσοντας ε, μια ε, γεφυρωτή αν θέλετε, δηλαδή μια γενική σφαιρική εφαρμογή ε, εργαλείων για την πρόληψη. Δηλαδή όταν μιλάμε για την πειρατεία αναφερόμαστε και στην αποτελεσματικότητα της ε, αναπτυξιακής πολιτικής, την προσπάθεια για τη μείωση της στόχιας για διατήρηση της ειρήνης, πρόληψη συγκρούσεων και ζητήματα σταθερότητας. Εγώ εκπροσωπώ μια μονάδα η οποία εργάζεται υπό των ζητημάτων ασφαλείας ε, και κατά συνέπεια η δική μου ενημέρωση αφορά τα όσα έχουμε κάνει από τη δική μας πλευρά για την καταπολέμηση της πειρατείας μέσω συγκεκριμένων προγραμμάτων ειδικότερα διαμέσου του εργαλείου για την ε, ε, συνεισφορά προς την σταθερότητα και την ειρήνη. Ε, σύντομα όπως το λέμε, το εργαλείο για τη σταθερότητα, προκειμένου να δημιουργήσουμε μακροπρόθεσμα δομές σε διάφορα μέρη του κόσμου, όπως αναφέρθηκαν αυτά ήδη από τον προηγούμενο μιλητή, προκειμένου να ε, βελτιώσουμε την ασφάλεια στη θάλασσα. Άρα λοιπόν η δική μου ε, παρέμβαση αφορά ζητήματα ασφαλείας. Υπάρχουν και άλλες επιτυχίες προφανώς, αλλά αυτές θα καλυφθούν αλλού. Άρα λοιπόν η δική μας βασική αρχή δεν είναι μόνο το ψήφισμα το οποίο ανέφερα μόλις τώρα, αλλά και τα όσα αναφέρονται στο εργαλείο για την συνεισφορά στη σταθερότητα, δηλαδή και τις προτεραιότητες οι οποίες αναφέρονται στο λόγο instrument, στο εργαλείο, αλλά και η στρατηγική 2014-2020 στο πλαίσιο της οποίας εφαρμόζεται αυτό το εργαλείο και το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 2014-2017. Είναι σαφές ότι εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνουμε, μας ανατίθεται η ερμοδιότητα στο πλαίσιο αυτού του εγγράφου και ε, στο πλαίσιο ε, περιφερειακών ε, πολιτικών, όπως για παράδειγμα οθήκη χθε ό,τι αφορά το κόλπο της Γουινέας, να ξεκινήσουμε με τη συνεισφορά μας για την καταπολέμηση της πειρατείας. Αν λοιπόν τα ποσά που έχουμε ενδεικτικά στην περίοδο 2007-2013 26,5 ε, ε, εκατομμύρια ευρώ δαπανήθηκαν και στην περίοδο 2014-2017 ε, προβλέπονται 16,5 εκατομμύρια ευρώ ως δαπάνες. Σε αυτό το πλαίσιο είναι πολύ σημαντικό για όλους εμάς που είμαστε εδώ να έχουμε και αυτά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια των ε, επόμενων ετών στο πλαίσιο της μεθοσοπρόθεσμης αναθεώρησης 2014-2017 προκειμένου να επαναληφθούν, δηλαδή να αναχρηματοδοτηθούν τα διάφορα ταμεία για την περίοδο 2018-2020. Και αυτό ε, βέβαια είναι σημαντικό γιατί υπάρχουν πολλές άλλες ε, ε προτεραιότητες οι οποίες ανταγωνίζονται τροποντινά αυτόν τον ε, τομέα. Ε, κατά κάποιο τρόπο λοιπόν είμαστε τυχεροί αν γιατί στο ανατολικό τμήμα της Αφρικής στο πλαίσιο του κώδικα διοντολογίας του Τζιμπουτή υπάρχει μια πολιτική όθηση, μια βούληση και αυτό που προσπαθούμε εμείς να κάνουμε σε εταιρική ε, βάση είναι να ε, συντονίσουμε τις διάφορες δράσεις οι οποίες ε, ε, λαμβάνουν χώρο στο πλαίσιο και να ενταχθούν στο πλαίσιο αυτού του κώδικα δεοντολογίας. Προσπαθούμε δηλαδή να έχουμε ένα περιφερειακό κέντρο συντονισμού στο Τζιμπουτί. Διεξάγουμε μία σειρά από εκπαιδευτικές δράσεις από την πλευρά των διαφόρων εκπροσώπων από τις χώρες που συμμετέχουν, αλλά ταυτόχρονα προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ή να οργανώσουμε διάφορες δράσεις στο πλαίσιο της επιβολής του νόμου. Εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα μαζί με την Interpol για την καλύτερη επιβολή του νόμου σε μία σειρά από χώρε προκειμένου να συμβάλλουμε στην καταστροφή, αν θέλετε, στην εξάλληψη των δικτύων πειρατεία και έχουμε ξεκινήσει τι εργασίε μα στον ευρύτερο ωκεανό. Δηλαδή προσπαθούμε εδώ να ε, συνδέσουμε τις διάφορους επιμέρους ε, περιοχές ε, του Ινδικού ωκεανού μέσω και πάλι κέντρων συντονισμού και εκπαίδευση, γιατί βέβαια είναι πολύ σημαντική και η εκπαίδευση στο πλαίσιο και της, του να αντιληφθούμε το τι ακριβώς συμβαίνει σε κάθε περιοχή. Τέλος, στον κόρπο τη γωνίας συμμερίζομαι πλήρως την αξιολόγηση που ακούσαμε μόλις τώρα από του συναδέλφου, Δηλαδή πραγματικά βλέπουμε μια μετατόπιση τη δραστηριότητα τη πειρατεία από την Ανατολική προ την Δυτική Αφρική. Ε, και κυρίω εδώ μιλάμε για αγροπή πετρελαίου ειδικότερα από πετρελοφόρα και Ε, έχουμε και μία σύνδεση των δραστηριοτήτων σε σχέση με τα όσα είχαν συμφωνηθεί και από τους ε, ηθήνοντες στο πλαίσιο του κώδικα δεντρολογίας του Ιαούντε. Όλα αυτά λοιπόν ε, μας δημιουργούν να δημιουργήσουμε ένα διαπεριφερειακό κέντρο συντονισμού. Έχουμε εμπειρογνώμονες εκεί επιτόπου και συνεχίζουμε και τις εκπαιδευτικές δράσεις. Αυτά λοιπόν εν ολίγης ως επισκόπηση των όσων κάνουμε στο πλαίσιο του εργαλείου για τη συνεισφορά σταθερότητα και την ειρήνη για την καταπολέμηση της πειρατείας. Ε, μιλάμε βέβαια ε, για ένα, ε, μια λύση αν θέλετε τελευταία ανάγκης, δηλαδή βράχη πρόθεσμη, ενώ στο επίπεδο της ΔΕΦΚΟ έχουμε την πιο μακροπρόθεσμη στρατηγική, δηλαδή δημιουργούμε τις δομές με αυτές τις χρηματοδοτήσεις οι οποίες θα μας επιτρέψουν την καταπολέμηση της πειρατείας, αναγνωρίζοντας βέβαια ότι πολλά θα πρέπει να γίνουν, ταυτόχρονα πρέπει να λαμβάνουν χώρο και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Γκάλερ πρώτος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριοι, σας ευχαριστώ για τις τοποθετήσεις σας. Περιμένω να φορέσετε τα ακουστικά σας. Είναι σημαντικό εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις αυτές με σύνολο μέτρων. Γνωρίζουμε αφενός ότι τα αίτια που οδηγούν στην πειρατεία συνήθως είναι εγχώρια. Από την άλλη μεριά πρέπει να είμαστε σε θέση να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας με την έννοια δηλαδή ότι υπερασπιζόμαστε τον εμπορικό μας στόλο που δραστηριοποιείται, που κυκλοφορεί στις θάλασσες ανατολικά και δυτικά της Αφρικής. Να μπορούμε να προστατεύσουμε τα σκάφη αυτά και με δημιουργία δικτύων όσων έχουν κοινά συμφέροντα. Ερώτηση. Πώς, τι επαφές έχετε, πώς δικτυώνεστε εσείς με την ίδια την αυτιλία, δηλαδή τι είδους πληροφορίες ανταλλάσσετε. Ο ίδιος εγώ προσωπικά έχω έρθει σε επαφή με μια οργάνωση που λέγεται OCIMF, τα αρχικά αυτά, εν δηλαδή, με έναν πλοίαρχο Κοτρέλ Η οργάνωση αυτή έχει αναπτύξει δίκτυα μέσω των οποίων ενημερώνει τα μέλη της, τους πλοιάρχους δηλαδή των πλοίων της, για την κατάσταση όπως αυτή διαμορφώνεται και συνεργάζονται μαζί τους. Και εμείς να συνεργαστούμε μαζί τους. Με ποιο τρόπο γίνεται αυτό. Εντάσσεται αυτό έτσι και αλλιώς στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας ή είναι περισσότερο τυχαίες οι επαφές αυτές. Και πιο συγκεκριμένη ερώτηση, χθες φαίνεται πως συνήλθε το Political Security Committee για τον κόλπο της Γουινέας. Έγινε αυτή η συνεδρίαση χθες. Βλέπω ότι νεύεται καταφατικά εσείς κύριε πρόσωπε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορείτε να πείτε κάτι πιο συγκεκριμένο για το τι συζητήθηκε η Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Η κυρία Άννα Γκόμης. Σας ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις που ήταν πολύ χρήσιμες. Νομίζω ότι επί του θέματος αυτού θα πρέπει να έχουμε και κάποιους εκπροσώπους ε, του αμυντικού κλάδου, στρατιωτικούς, που να έχουν εμπλακεί διότι η εμπειρία τους είναι πολύ χρήσιμη ώστε να καταλάβουμε πώς αυτά τα δεδομένα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην ε, Δυτική Αφρική διότι υπήρξε και αυτή η μετατόπιση από την Ανατολική προς τη Δυτική Αφρική όπως καταλάβαμε όπως και εμπειρογνώμονες ε, ακαθημαϊκοί εγώ πέρυσι ήμουνα στο Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, στο μέση του Ατλαντικού, σε ένα εργαστήριο που είχε διοργανώσει η Βρετανική κυβέρνηση, όπου είχαμε και μία μελέτη από το Βασιλικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών, σχετικά ακριβώς με τα αυξανόμενα κρούσματα πειρατεία στην Δυτική Αφρική, την φύση δηλαδή των εγκληματικών αυτών δραστηριοτήτων. Πολλά από αυτά έχουν σχέση με το πετρέλαιο και στην Ιγυρία αλλά και με το παράνομο εμπόριο όπλων και ναρκωτικών και από ό,τι φαίνεται πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ενέχονται. Το επαναλαμβάνω, πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ναυτιλιακών, και άλλων κλάδων ενέχονται, εμπλέκονται. Υπήρξε μια περίπτωση σουηδικής εταιρείας Stene Oil που ήταν υπεύθυνη για σκάφη που μετέφεραν πετρέλαιο που είχε κλαπεί στην Ιγυρία ή στα ύδατα που ήταν στον έλεγχο του Σαοτομέ και μετέφεραν το πετρέλαιο από μικρότερα σκάφη σε μεγαλύτερα και πλέον νομιμοποιημένα νόμιμα σκάφη στη μεταφόρτωση μέσω μαλτέζικων ε, ε, επιχειρήσεων. Καθότι βεβαίως το ελαχιστότατο, το, το πολύ περιορισμένο ναυτικό της μικρής αυτής χώρας έκανε ό,τι μπορούσε και συνέλαβε τους ε, πλοιάρχους ε, τους δύο. Ε, έχει γίνει μία δίωξη τώρα που εκδικάζεται στο Αμβούργο και έχουν ασκήσει οι επιχειρήσεις, αυτοί, οι επιχειρήσεις αυτές μήνυση κατά της χώρας αυτής που έκανε αυτά που έπρεπε. Και μιλούμε για μια χώρα που είναι και μέλος της ACP ΑΚΕ. Και θα ήθελα να ξέρω τι κάνουμε ακριβώς για να βοηθήσουμε χώρες που θέλουν να καταπολεμήσουν τα φαινόμενα αυτά και που δεν έχουν τα μέσα στη διάθεσή τους. Και δεν πρόκειται για μεμονωμένες προσπάθειες χωρών όπως η Πορτογαλία, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο που έχουν δεσμούς με τέτοιες χώρες, αλλά πρέπει να είναι ρόλος και για την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως και για τις Ηνωμένε Πολιτείε που είχαμε εκπροσώπηση ε, στο σεμινάριο εκείνο στο Σάτομε. Είχαμε δύο εργαστήρια, ένα ε, διοργανωμένο από τους Βρετανούς και ένα από τους Αμερικανούς. Νομίζω λοιπόν ότι αυτά τα φαινόμενα είναι ήδη πολύ σοβαρά και γίνονται πιο σοβαρά ακόμα. Όπως μας είπαν και τα μέλη του πάνελ, αλλά και γιατί σύντομα θα έχει ολοκληρωθεί η διεύρυνση της διόρυχας του Παναμά με πολύ σημαντικό αντίκτυπο για την αύξηση των κρουσμάτων λαθρεμπορίου στον κόλπο της Γουινέας αύξηση και του νομίμου και του παράνομου εμπορίου δηλαδή και οι λαθρέμποροι ναρκωτικών ε, χρησιμοποιούν πλέον και υποβρύχια είναι όλο και πιο συζητημένοι στις μεθόδους τους δεν μπορούμε λοιπόν να αρκούμεθα ε, με την αποτύπωση της αλλαγής της τάσης, της γεωγραφικής, πρέπει να είμαστε προδραστικοί, πριν να προλαμβάνουμε τα γεγονότα αυτά, τα φαινόμενα αυτά και ποια μέσα χρειάζονται με τους εταίρους μας, τους περιφερειακούς, ώστε να επιτύχουμε υποστήριξη όχι μόνο από ιδιωτικές ε, οργανώσεις ε, που συνδέονται, όπως είπε και ο συνάδελφος, με την ε, ναυτιλία, αλλά τι κάνουμε για να ενισχύσουμε τις αρχές των χωρών της περιοχής, των περιοχών αυτών. Μιλούμε για κατάρτιση ε, των, ε, του προσωπικού, των σκαφών, την χαρτογράφηση των όποιων εγκαταστάσεων έχουμε στη θέση μας. για παράδειγμα οι βάσεις ε, στις Αζόρες που αυτή τη στιγμή εν μέρει εγκαταλείπουν οι Αμερικανοί για να πω ένα παράδειγμα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ωραιότατα ως κέντρα παρατήρησης, ε, επιτήρησης, περιπολιών οι άλλες ε, εγκαταστάσεις στο Κάμπο Βέρντι, στο Σατομέ, στην Αγκόλα, σε άλλες χώρες που θα μπορούσαν να ενδιαφέρονται και να είναι διαθέσιμες για μια τέτοια προσπάθεια. Και βεβαίως για την ε, δικαστική προσπάθεια. Γιατί ε, ώστε να αποφεύγουμε δηλαδή τέτοια φαινόμενα ε, προσφυγή σε ιδιωτικά δικαστήρια τα οποία είναι λίγο δύσκολο να αντιμετωπίζονται. Και θα ήθελα να ρωτήσω τους εμπειρογνώμονες πώς βλέπουν την διασύνδεση με τον αυξανόμενο κίνδυνο τρομοκρατίας που δεν περιορίζεται μόνο στη γη, στις χερσαίες επιχειρήσεις, στο, Μα, στο Μαλί, στην Ιγυρία, τον Μπόκο Χαράμ και αυτό σχετίζεται πάρα πολύ η δραστηριότητά του με το πετρέλαιο προφανώς. Πώς προετοιμαζόμαστε δηλαδή και πώς προσπαθούμε να προλάβουμε αυτή την απειλή με τα μαθήματα της Ανατολικής Αφρικής και της ε, Αταλάντα κυρίες. Σας ευχαριστώ. Α, και μία τελευταία ερώτηση. Ζητώ συγγνώμη, Πρόεδρε. Μία τελευταία ερώτηση. Όταν έκανα την μελέτη για την θαλάσσια διάσταση της ESTP, βρήκα τη ΕΜΣΑ, ο οργανισμός αυτός που βασίζεται στη Λισαβόνα, για την ασφάλεια στη θάλασσα προκειμένου να εξασφαλίσει ακριβώς ασφάλεια για τους θαλασσοπόρους, ασφάλεια για περιβαλλοντικές και άλλες καταστροφές. Είχε τα μέσα, αλλά δεν είχε την εντολή. Δεν είχε την εντολή ε, να προβαίνει σε υποστήριξη ε, επιχειρήσεων όπως η Αταλάντα ή άλλων παρεμφερών προκειμένου να αντιμετωπίσουμε απειλές όπως η πειρατεία και άλλες. Αυτό το έκαναν στην ουσία, αλλά εκτός εντολής, το οποίο είναι γελίο, απολύτως. Ήθελα να σας ρωτήσω αν αυτό έχει αλλάξει και αν αναγνωρίζομαι, επιτέλους, ότι η ΕΜΣΑ έχει αυτό το δυναμικό, έχει αυτές τις δυνατότητες και μπορεί και νομικά και νομίμως και ανοιχτά να συνεργαστεί μαζί μας για τέτοια θέματα. Thank you, madam. Mr. Ευχαριστούμε, ο κύριος Τουνακέλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα ε, να σας ευχαριστήσω για μια πολύ χρήσιμη και ε, σφαιρική παρουσίαση της ε, κατάστασης. Όπως είπαμε, όπως αναφέρατε και εσείς, τα τελευταία χρόνια η βασική κατάσταση δεν έχει αλλάξει, βασικές παράμετροι αλλά έχει βελτιωθεί κάπως και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Βαντερμέλ σε σχέση με τις πληροφορίες που μας έδωσε, δηλαδή σε ό,τι αφορά ε, τις εργασίες που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με αυτό το ζήτημα στη Σομαλία. Ε, όμως ε, στο, το ερώτημά μου είναι η UNODC και το, η ομάδα επαφής ε, πράγματι έχουν καταφέρει να έχουν μια καλή επικοινωνία μεταξύ τους και το κύριο ζητούμενο ήταν να αναγνωριστούν οι κρίσιμες ε, ανάγκες και η κάλυψή τους ε, σε έστω χρονικό διάστημα. Όμως αναφέρεται επίσης ότι μια απόλυτη προϋπόθεση είναι μια, ένας πολιετής και πλήρης σχεδιασμός. Θα ήθελα ε, λοιπόν να σας ρωτήσω ποια, ε, ποιες είναι οι προοπτικές μα ώστε να επιτύχουμε ένα τέτοιο μακροπρόθεσμο και γενικό σχεδιασμό. Επίσης αναφέρεται ότι έγιναν κάποιες ε, προτάσεις να διοργανωθεί μια αποστολή των ε, ΗΠΑ ώστε να υπάρχουν δηλαδή ένοπλες ε, ομάδες εν πλώ επάνω σε αυτά τα πλοία. Το δικό μου ερώτημα είναι υπάρχουν μία σειρά από ομάδες ε, ασφαλείας ε, και αντιτρομοκρατές που ήδη δραστηριοποιούνται και βρίσκονται δηλαδή πάνω σε αυτά τα πλοία ε, που έχουν δημιουργηθεί μέσω διμερών συμφωνιών ή που βρίσκονται πάνω σε ειδικά διαμορφωμένα πλοία καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι το νομικό πλαίσιο. Πού εντάσσονται δηλαδή τέτοιου είδους ομάδες. γιατί οι δραστηριότητε του έχουν δημιουργήσει κάποια προβλήματα με τι γειτονικέ χώρες όπως η Ινδία. Υπήρχε δηλαδή η περίπτωση των δύο Ιταλών ε, των οποίοι ήταν, κρατούμενοι στην Ινδία. Υπήρχε μετά η περίπτωση 14 πολιτών της Αστωνίας και 6 πολίτες ε, των, ε, του Ηνωμένου Βασιλείου που κρατούνται στην Ινδία από το 2013 χωρίς να τους έχουν απαντηληθεί επίσημες κατηγορίες ή έχουν αδωθεί σε ό,τι αφορά ενδεχόμενε παραβιάσεις της ελληνικής νομοθεσίας, αλλά παρόλα αυτά αυτοί οι ε, πολίτες παραμένουν κρατούμενοι στην Ινδία και ε, κ. Μογκερίνη έχει ε, κάνει κάποια Μογκερίνη έχει κάνει κάποιες σημαντικές προσπάθειες ούτως ώστε να απελευθερωθούν αυτά τα άτομα. Οπότε το δικό μας ερώτημα είναι χρειαζόμαστε ένα σαφέστερο νομικό πλαίσιο ε, για αυτές τις περιπτώσεις και προκειμένου να προστατεύσουμε καλύτερα τα δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τέτοιες περιπτώσεις. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Εάν δεν υπάρχουν άλλα ερωτήματα, θα ήθελα να αναφερθώ και πάλι ε, στη Δυτική Αφρική και στον κόλπο της Γουινέας και να χαιρετήσω βέβαια και το ερώτημα του κυρίου Γκάλερ σε ό,τι αφορά δηλαδή το σχέδιο δράσης. Οπότε θα μπορούσαν ε, ομιλητές να μας διευκρινίσουν λίγο ε, το πώς έχει γίνει αυτή η μετατόπιση της ε, δραστηριότητας ε, προς την Δυτική Αφρική και το ποιες, ποια δράση θα πρέπει να αναλάβουν τα διάφορα θεσμικά όργανα ώστε να εφαρμοστούν και σχετικά προγράμματα. Γιατί είναι σαφές πως δεν έχουμε εδώ να κάνουμε μόνο με πειρατεία. Συμφωνώ με αυτό δηλαδή που είπατε ότι εδώ αποτελεί τον τελευταίο κρίκο μιας ολόκληρης αλυσίδας στο φαινόμενο της πειρατείας και κατά συνέπεια μπορεί, ε, αποτελεί δηλαδή τον σύνδεσμο προς άλλες δραστηριότητες οι οποίες είναι ακόμα πιο επικίνδυνες. Ε, θεωρείτε πως αυτό το φαινόμενο για παράδειγμα της ε, μετατόπισης πειρατείας σχετίζεται και με την αυξημένη δραστηριότητα ακραίων οργανώσεων όπως για παράδειγμα η Μπόκο Χαράμ, ενδεχομένως η υπάρχει ένα δρομολόγιο από την Βενεζουέλα που πάει προς την Δυτική Αφρική, ένας διάβλος δηλαδή λαθεμπορίων ναρκωτικών και είμαι βέβαια πως υπάρχουν και άλλα τέτοιες, άλλες τέτοιες ε, ε, διάβλη δρομολόγια, αν θέλετε, οργανωμένου εγκλήματο. Ε, τι θα πρέπει να κάνουμε εμεί σε αυτή την περίπτωση, πώ πρέπει να συντονίσουμε τι δράσει μα, ώστε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά αυτά τα προβλήματα. Έχεις το λόγο. Uh, uh, thank you very much for the uh, um, interventions which some very interesting. Σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας. Να αναφερθώ πρώτα στα θέματα συνεργασίας. Είναι αλήθεια ότι η συνεργασία μεταξύ εκπροσώπων των στρατιωτικών του κλάδου και των κυβερνητικών φορέων είναι μια απόδειξη της αποτελεσματικότητας της ε, ομάδας επαφής και του μηχανισμού του Μπαχρέιν που συνομαδοποίησε κατά αντίστοιχο τρόπο τις ναυτικές ε, τους ναυτικούς ενδιαφερόμενους φορείς των πολεμικών ναυτικών δηλαδή είναι σίγουρα αλήθεια για να στραφώ καταρχάς στην Ανατολική Αφρική ότι βλέπουμε μια διαφοροποίηση στις τάσεις της εγκληματικότητας στη θάλασσα και στο λαθρεμπόριο και στην εμπορία ανθρώπων και οι άνθρωποι που έχουν παράνομα έσοδα δεν είναι από τις δραστηριότητες αυτές δεν είναι αυτοί που έχουμε ήδη κρατούμενους και για να αναλάβω την ηρωίνη ως παράδειγμα ο πόλεμος στη Συρία και οι ενισχυμένες προσπάθειες ε, ε, στην Κεντρική Αφρική, η Τανζανία, περιορισμού των οδών αυτών, έχει προκαλέσει μία καμπή, μία μεταστροφή ε, στον τρόπο με τον οποίο επιχειρούν οι οργανώσεις αυτές στις θαλάσσιες οδούς. και λόγω της νομοθεσίας συγκεκριμένων χωρών υπάρχουν ελκυστικές αν θέλετε ζώνες για τη δράση των εγκληματικών αυτών ομάδων. Αναφερθήκατε επίσης τα ε, στα θέματα της τρομοκρατίας. Έχουμε ε, το ψήφισμα 2985 των Ηνωμένων Αθηνών ακριβώς για το σχετισμό αυτό και εδώ για παράδειγμα οι Ταλιμπάν έχουν σημαντικά έσοδα από το λαθρεμπόριο του Ινδικού ωκεανού. Η al κυρίως από το λαθρεμπόριο ε, άνθρακα κάρβουνου και άλλα αντίστοιχα τέτοια κρούσματα. Ε, Επίση μας ρωτήσατε σχετικά με το σχεδιασμό, τον πλήρη σχεδιασμό ε, σε σχέση με τη Σομαλία μέσω του μηχανισμού Compact, ε, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και βασικός αρχιτέκτον αν θέλετε, για, την, για το συντονισμό της ανταπόκρισης αυτής και για τα θέματα της ασφάλειας το τελευταίο που αναφέρατε. Είναι τεράστια πρόκληση επί τη βάση τη νομική. Εγώ προέρχομαι από τις νομικές υπηρεσίες του πολεμικού ναυτικού και είναι κυρίως ευθύνη της ε, χώρας σημαίας. Ε, έχουμε πολλές περιπτώσεις ε, σημαίων ευκαιρίας και χώρες που δεν αναλαμβάνουν κανένας είδους ευθύνη για όλα αυτά. Και αν δεχθεί ένας κάπως μια επίθεση από πειρατέ, η πρώτη ευθύνη και για τους όποιους ομήρους ή την ε, ένοπλο ανταπόκριση κτλ. Ε, είναι της ε, χώρας σημαίας. Αλλά βλέπουμε ότι καμία από τις χώρες αυτές σημειών ευκαιρίας δεν έχει ενδιαφερθεί να ασχοληθεί με τη διαχείριση των θεμάτων αυτών, τους ομήρους, την πολεμική επιχείρηση εφόσον χρειαστεί, έχουν απολύτως παρετηθεί στις, ε, στους διεθνείς φορείς, στο ναυτικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπόλοιπων εταίρων που επιχειρούν στις ζώνες αυτές τις προβληματικές και επομένως θα έπρεπε κανεί να καταλήξει το συμπέρασμα ότι δεν θα έπρεπε να δέχεται υπηρεσίε τόσο χαμηλής ποιότητας για να το ονομάσω έτσι από τις χώρες αυτές που προσφέρουν τη σημαία τους με τόσο εύκολο τρόπο και επιφανειακό. Όλα λοιπόν ε, αφήνονται στις, στους ε, τοπικούς φορείς, στους τοπικούς λιμένες, εκεί που έχει γίνει οποιαδήποτε μεταφόρτωση. Έχουμε δει για παραδείγματα στην Ινδία, για παράδειγμα, ε, και είναι πολύ σημαντικό το θέμα της κατάρτισης των φρουρών των σκαφών. Έχουμε ιδιωτικές επιχειρήσεις ε, ακριβώς που ασχολούνται με τα θέματα αυτά ε, στις μεταφορές και στη Σομαλία και σε άλλες περιοχές. Ας δώσω όμως λίγο χρόνο και στα υπόλοιπα μέλη του πάνελ. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπατε για τη σημαίες ευκαιρίας Εσείς κύριε Χούμπεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να συμπληρώσω αυτά που είπε ο Άλαν και ας αρχίσω με την ερώτηση του κύριου Γκάλερ για την ροή πληροφοριών από την εμπορική ναυτιλία. Θα γνωρίζετε ότι μέσα στα πλαίσια της επιχείρησης Αταλάντη δημιουργήθηκε και ένα επιχειρησιακό κέντρο για την περιοχή. Είναι ένα κέντρο συγκέντρωση των πληροφοριών όπου οι... τα εμπορικά καράβια δηλώνουν ποια διαδρομή θα ακολουθήσουν μέσα από τα επικίνδυνα ύδατα. Και όταν επιστρέφουν κάνουν μια αξιολόγηση του κινδύνου και κυρίως διασφαλίζουν ότι κάποιος τα προσέχει τα σκάφια αυτά. Υπάρχουν και άλλα δύο κέντρα τα οποία παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες. Η Maritime Trade Organization και το NATO Shipping Center. UKMTO και NATO Shipping Center έχουν παγκόσμιο πλαίσιο αρμοδιοτήτων. Το USMCO έχει σχέση μόνο με την Αταλάντη και μόνο με τη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή. Το πολιτικό θέμα που καλούνται να απαντήσουν οι χώρες μέλη είναι όταν θα αρχίσουν να επανεξετάζουν την εντολή και ίσως τον τερματισμό της εντολής της Αταλάντης, το Maritime Security Center θα πρέπει και αυτό να σταματήσει τις δραστηριότητε του. Για την ώρα όμως το feedback που λαμβάνουμε είναι ότι οι υπηρεσίες που προσφέρει το κέντρο αυτό στην ναυτιλία έχουν τόσο μεγάλη αξία που η ερώτηση μάλλον θα πρέπει να είναι αν θα πρέπει να παραταθεί η εντολή του για SMCO και να καλύψει ολόκληρη την Αφρική και, την, ε, τον κόλπο της Γουινέας. Είναι πολιτικό το θέμα βέβαια, το οποίο θα κληθούν να απαντήσουν οι χώρες μέλη. Ίσως επίσης ακούσατε τις προφορίες από τους αδέρφους της ΟΚΕΜΦ ότι ο κλάδος φτιάχνει δικό του εντός εισαγωγικών δικά του κέντρα στον κόλπο της Γουινέας για την εμπορική ναυτιλία είναι ζήτημα εμπιστοσύνη Να μοιραστούν τι πληροφορίε αυτέ, δηλαδή μαζί μα. Για παράδειγμα δεδομένα GPS των πλοίων, διότι δεν θέλουν να είναι γνωστά αυτά τα πράγματα, ούτε και βεβαίω να δημοσιεύονται στο διαδίκτυο. Αν μπορούν λοιπόν να λειτουργήσουν, να κάνουν business με τον εταίρο αυτόν. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το κέντρο αυτό μέσα στα πλαίσια της επιχείρησης Αταλάντη και έχει τώρα χέρι εμπιστοσύνη. Από αυτά που έχω καταλάβει από τι επαφέ μου με τον κλάδο τη εμπορική ναυτιλία, η εμπιστοσύνη ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί με τα κέντρα παροχή πληροφοριών για τον κόλπο τη Γουινέα. Είναι λοιπόν μακροπρόθεσμη προσπάθεια αυτή που θα πρέπει να γίνει πριν να αποκατασταθεί αυτό ο αξιόπιστος σύνδεσμο μεταξύ των ε, επιχειρήσεων και, το, και του κέντρου αυτού. Τώρα, απαντώντας σε ορισμένε άλλε ερωτήσει που έθεσε η κυρία Γκόμης, για τη γενική αναστάτωση που βλέπουμε στον χώρο της ναυτιλίας. Μιλήσατε και για, το, για τη διόρυγα του Παναμά. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω μια έκφραση του William Νάλοριτζ. Μίλησε για την θάλασσα των παρανόμων, δείχνοντας μια κατάσταση που λέει ότι δεν υπάρχει επαρκής διακυβέρνηση ούτε και επαρκής πόρη για να διακυβέρνηση τη τεράστια αυτής της περιοχής των θαλασσών. Βλέπουμε επίσης πολλές από τις προκλήσεις αυτές να αλληλοενισχύονται και ιδίω αυτό είναι εμφανές και οξύ όταν έχουμε αυτό τον ενδεχόμενο σύνδεσμο μεταξύ της πειρατείας ως ναυτικού εγκλήματος δηλαδή συλλογής πόρων και της δημοκρατίας. Και από στρατηγική αλλά και από άποψη συλλογή πληροφοριών και ασφάλειας πρέπει να επαγρυπνούμε απολύτως και να παρατηρούμε την εξέλιξη του φαινομένου. Επανέρχομαι στο Contact Group, που, Contact Group 5 όπου ηγείται η Ιταλία. Υπάρχει λοιπόν η παρακολούθηση των ροών που βρέχονται από την πειρατεία και ενδιαφέρονται ιδίω να στοχεύσουν στους εγκεφάλους πίσω από την ε, υπόθεση αυτή. Για παράδειγμα, εγκέφαλοι στο Ντουμπάι, οι οποίοι κατευθύνουν τα νήματα και χρηματοδοτούν τις επιχειρήσεις αυτές της πειρατείας. Να εντοπίζουν λοιπόν χώρα η οποία θα είναι διατεθειμένη να φέρει την υπόθεση στο δικαστήριο, να προσφέρουν πληροφορίες ώστε να είναι ισχυρή η θέση της χώρας απέναντι στο δικαστήριο, στην υπόθεση αυτή δηλαδή. Και αυτό μπορεί να επαναληφθεί και σε άλλους τομείς. Κυρία Γκόμες, μιλήσατε για την ΕΜΣΑ, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θαλάσσιας Ασφάλειας. Υπάρχει και το κέντρο των δορυφόρων, Satellite Center, Αυτό μέσα στο πλαίσιο της συνολικής ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ασφάλεια στις θάλασσες που έχει εντοπίσει πώς διαμορφώνονται οι διάφορες σχέσεις και στήριξη που μπορούν να δώσουν οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί σε αποστολές της CSDP. Μπορούν να ενισχυθούν αυτά. Και η διοδόση θα πρέπει να γίνει με χρήση σωστών διαδικασιών, επομένως με αλλαγή της επίσημης εντολής των οργανισμών αυτών. Όμως έχει εντοπιστεί το θέμα και προχωρεί, θα χρειαστεί χρόνο, αλλά βέβαια η διεύρυνση της εντολής της ΕΜΣΑ για μας είναι κάτι το απόλυτα αναγκαίο. Τέλος, απαντώ στον κύριο Κέλαμ. Το Multi-Year Comprehensive Planning, αυτός ο σε βάθος σχεδιασμός, πολιτή σε βάθος σχεδιασμός. Βεβαίως αυτό είναι το Άγιο Δισκοπότηρο για μας. Χρειαζόμαστε ένα διεθνές περιβάλλον με εκπροσώπους κρατικών οργανισμών, κρατικών αρχών, αλλά και του ιδιωτικού τομέα. Αυτό είναι δύσκολο να επιτευχθεί και ποτέ δεν θα υπάρξει μια ενιαία αρχή σχεδιασμού που να είναι υπεύθυνη για αυτό τον πολιετή σχεδιασμό. Το μόνο πράγμα λοιπόν που μπορεί να γίνει και το καλύτερο που μπορούμε να επιτύχουμε είναι να εξασφαλίσουμε ορατότητα για όλα αυτά τα άλλα ενδιαφερόμενα μενή, stakeholder, και να δείξουμε ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο σε εθελοντική βάση. Αυτό είναι και το νόημα της παρέμβασής μου να σας εξηγήσω ποια είναι η εμπειρία δηλαδή της ομάδας επαφών, ότι αυτό το βήμα είναι καλό για να προσεγγίσουν αυτές οι διαφορετικές ομάδες ενδιαφερομένων, η μεν της δε, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για να υπάρξει αυτή η διαρκή στη βιώσιμη απάντηση σε ένα πάρα πολύ περίπλοκο πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ κύριε ε, Χούμπεν. Ο κύριος Βάντερ Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για τα ερωτήματα που θέσατε ε, και τα οποία πράγματι έθεσαν σε ένα γενικότερο πλαίσιο τα ζητήματα που συζητάμε εδώ. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε και εμείς το πλαίσιο του σχεδίου δράσης για, για τον κόλπο της Γουινέα, το οποίο θετήθηκε χθες από το Συμβούλιο. Ο ένα από τους συντάκτες αυτού του κειμένου είναι εδώ. που συμμετείχε στην σύνταξη του κειμένου είναι σαφές λοιπόν σε αυτήν την ε, στρατηγική και σε αυτό το σχέδιο δράσης βλέπουμε τώρα για πρώτη πλέον φορά την εφαρμογή της ολικής ε, προσέγγισης της υπηρεσίας της ε, εξωτερικής σχέσης σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη αυτή περιοχή. Ε, και αυτό, αυτή ακριβώς η προσέγγιση αφορά όλα αυτά τα ζητήματα που θέσατε πρόεδρε, δηλαδή την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, το ζήτημα της αυτιλιακής ασφάλειας, της ασφάλειας στη θάλασσα και ζητήματα επιβολής του νόμου σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και υπογραμμίζοντας ε, ταυτόχρονα ε, την ε, κατάσταση, την οικονομική κατάσταση σε αυτές τις χώρες και την προώθηση ενός ασφαλούς ναυτιλιακού τομέα. Άρα λοιπόν αυτό που βλέπουμε στο λόγο έγγραφο είναι όχι μόνο η σύνδεση με τα όσα έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας, της πρόληψης συγκρούσεων και ούτω καθεξής, αλλά και με όλα όσα εκείνα προσπαθήσαμε να κάνουμε στο πλαίσιο του ε, εργαλείου για την σταθερότητα και την ε, ειρήνη. Το σχέδιο δράσης επίσης ονοματίζει ε, συγκεκριμένες δράσεις ανάλογα με την κλίμακα ε, της απειλής ε, αναφέρει το μίσος ο οποίος θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε για την καλύτερη συνεργασία τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διεθνές επίπεδο αλλά και δράσεις για μια καλή οικονομική ανάπτυξη ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις παράκτης κοινότητες και βέβαια προς όφελος της ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας. Ε, κυρία Πρόεδρε, καθημερινά ε, και εμεί έχουμε ενώπιον μα διάφορε ανταγωνιστικέ μεταξύ του, αν θέλετε, προτεραιότητε στο πλαίσιο του ίδιου εργαλείου. Έχουμε καταπολέμηση τη τρομοκρατία, έχουμε καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο ε, και έχουμε ταυτόχρονα προστασία τη κρίσιμη υποδομή. Ε, τα ζητήματα λοιπόν τη αυτιλική ασφάλεια καλύπτονται στο πλαίσιο της προστασίας των κρίσιμων φυλακών ε, υποδομών γιατί γνωρίζουμε ότι εδώ υπάρχουν πολύ σημαντικά ε, συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, τα οποία αφορούν ακριβώς την ασφαλή διέλευση των δικών μας ναυτών διαμέσου αυτών των περιοχών. Ναι, υπάρχουν πολλά μεγάλα προγράμματα τα οποία δημιουργούνται ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση. Σήμερα, για παράδειγμα, είναι επίκαιρο το ζήτημα τη ε, πειρατεία. Και αυτό που προσπαθούμε εμεί να κάνουμε κάθε φορά είναι να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένε ε, πτυχέ που σχετίζονται με αυτέ τι εγκληματικέ δραστηριότητε. Δηλαδή, διασφαλίζουμε ότι έχουμε συγκεκριμένε δομέ για την αντιμετώπιση ε, των εν λόγω ζητημάτων. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά ειδικότερα την πτυχή του οργανωμένου εγκλήματο. Μέσω διακυβέρνηση στις συγκεκριμένες ε, χώρες μέσω ε, του να μάθουν οι χώρες να συνεργάζονται μεταξύ τους ε, και σε εσωτερικό αλλά και σε εξωτερικό επίπεδο, σε περιφερειακό για παράδειγμα επίπεδο, όπως είδαμε στην κρίση του έμπολα, αναγνωρίστηκε ότι υπάρχει μια σημαντική ανάγκη για ε, συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών, των αρμοδίων υπηρεσιών, αλλά και διασυνοριακή συνεργασία. Άρα λοιπόν αυτή είναι η δική μου άποψη. Επί της ουσίας, μακροπρόθεσμα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε τις δομές που χρειαζόμαστε, τα εργαλεία εκείνα που χρειαζόμαστε σε αυτές τις χώρες, στο πλαίσιο ε, της καταπολέμησης αυτών των φαινομένων, αν θέλετε, που αποτελούν την ε, αρνητική τυχή της παγκοσμιοποίησης. Είναι εύκολο αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Όχι. Είναι, έχουμε μεγάλες δυσκολίες, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την εξέβρεση των ε, σωστών ε, εταίρων, τη δημιουργία των ε, focal points, συνεργασίας μέσω των οργανώσεων. Και στο πλαίσιο, για παράδειγμα, που αναφέρθηκε το πολύ σημαντικό ζήτημα της συνεργασίας στον κόλπο της Γουινέας. Θέλουμε να συνεργαζόμαστε με τις περιφερειακές οργανώσεις όπως την ΕΚΟΣ και άλλες γιατί είναι σημαντική η εταίρη και θεωρούμε ότι τα εν λόγω ζητήματα δεν μπορούν να επιληθούν σε εθνικό επίπεδο. Χρειαζόμαστε περιφερειακή ή ακόμα και διαπεριφερειακή προσέγγιση. Αναφερόμαστε εθνικό και για παράδειγμα, ναι. Αυτό προσπαθεί να, να κάνουμε δηλαδή στο πλαίσιο αυτού του, του προγράμματο. Δηλαδή να δούμε το τι συμβαίνει στη Λατινική Αμερική, τι συμβαίνει στην Αφρική και σε όλε τι σχετικέ ε, περιοχέ έχουμε και ένα άλλο ε, πρόγραμμα ε, στο πλαίσιο για παράδειγμα τη νομολογία του Σκοκάνης για την ε, βελτίωση της ασφάλειας στα αεροδρόμια και επίσης ένα πρόγραμμα σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αστυνομικών αρχών και εμπλέκοντας και την Ευρωπόλ και την Ιντερπόλ. Ένα πρόγραμμα ράπης σύστημα δηλαδή αστυνομική συνεργασία στη Δυτική Αφρική. Είναι λοιπόν όλα αυτά δράσει τι οποίε ε, έχουμε θέσει σε εφαρμογή, αλλά εκείνο που είναι σημαντικό είναι να έχουμε και ταυτόχρονα εκπαίδευση ε, στι ε, κάθε χώρε, ούτω ώστε εκείνοι οι οποίοι συλλαμβάνονται πράγματι να έχουν και μια, να δικάζονται και να καταδικάζονται όπω πρέπει. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε μακροπρόθεσμα ε, δέσμευση της δικής μας δραστηριότητας. Χρειαζόμαστε τα σωστά εργαλεία, χρειαζόμαστε όμως και περιφερειακή συνεργασία, χρειαζόμαστε ε, την ε, κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας και εδώ θεωρούμε πως θα μπορέσουμε να επιτύχουμε σε αυτό το συγκεκριμένο τομέα επιτυχίες και στο μέλλον γνωρίζουμε πως ο ιδιωτικό τομέα έχει δημιουργήσει τα δικά του συστήματα αλλά δεν μπορούν να αποτελέσουν μια βιώσιμη αναλλακτική τα συστήματα αυτά των, ε, του ιδιωτικού τομέα. Οι ίδιε οι χώρε δηλαδή εμπλεκόμενε θα πρέπει να δημιουργήσουν τι δικέ του ε, δομέ. Αλλά και σε συνδυασμό με τα όσα συμβαίνουν στο επίπεδο του ιδιωτικού τομέα. Ε, ώστε να μην έχουμε δηλαδή την επανάληψη και αλληλεπικάλυψη των ίδιων εργασιών. Άρα λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο, δηλαδή σε αυτό το συνδυασμό τη καταπολέμηση τη δημοκρατία, τη ναυτιλιακή ασφάλεια, καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο, προσπαθούμε να χρηματοδοτήσουμε ε, το, ε, δράσεις όπως για παράδειγμα το, το κέντρο στο Αμπουδάμπι, η πρωτοβουλία στη Γενέβη, ούτω ώστε να επιτύχουμε τα όσα μπορούμε ε, να επιτύχουμε στο πλαίσιο της καταπολέμησης της δημοκρατίας με βάση τα όσα ε, από την πλευρά του Συμβουλίου το Φεβρουάριο. Αυτά λοιπόν από τη δική μας πλευρά αναμένουμε με ενδιαφέρον την ανταλλαγή απόψεων με εσά σε ό,τι αφορά αυτές τις προκλήσεις ε, και έχουμε δημιουργήσει ε, και μια ε, εκδήλωση του ώστε και ε, μέλη του Κοινοβουλίου να έρθουν να συζητήσουν με συναδέλφους και να δείτε κι εσείς από την πλευρά σας δηλαδή με βάση τη σας εμπειρία πώς μπορείτε να συνεισφέρετε σε αυτές τις δράσεις από την πλευρά πάλι την γωνία της ασφάλειας. Σας ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποια άλλη παρατήρηση. Αν δεν έχουμε θα ήθελα εδώ κάπου να ολοκληρώσουμε αυτή τη διήμερη συνάντηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη του πάνελ για τις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις και παρουσιάσεις τους. Θα παρακολουθήσουμε τις ε, εξέλιξεις και η επόμενη συνεδρίαση με αυτή τη θεματική σίγουρα φέτος θα διοργανωθεί προκειμένου να έχουμε μια στενή παρακολούθηση, ίσως να έχουμε και εκπροσώπηση του ιδιωτικού κλάδου σχετικά με τις δικές τους δυνατότητες ε, συνεισφορά στην προστασία του, του στόλου, των εμπορευμάτων και του προσωπικού ε, των κρατών μελών. Και εδώ θα ήθελα να υπογραμμίσω τις παρατηρήσεις του κυρίου Κόλ σχετικά με την αναγκαιότητα αποσαφήνισης του νομικού πλησίου των εμπορικών στόλων, διότι αυτή τη στιγμή υπό τα των εξελίξεων το καθεστώς στο οποίο κινούνται οι εμπορικοί στόλοι δεν μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τα προβλήματα και τις προκλήσεις. Σας ευχαριστώ λοιπόν και θα ήθελα να συγχαρώ και τον ΕΑΣ και άλλες ε, οργανώσεις, φορείς, οργανισμούς ε, σχετικά με τις προσπάθειες απελευθέρωσης ομήρων. Πρέπει να υποστηρίξουμε κάθε δράση προκειμένου να απελευθερωθούν και οι υπόλοιποι οι απομένοντες 26 όμοιροι. Και η Υποεπιτροπή Αμυντικών Θεμάτων οπωσδήποτε θα υποστήριζε οποιονδήποτε φορέα και οργανισμό ενέχεται σε μια τέτοια προσπάθεια. Ευχαριστώ λοιπόν όλους. Ε, στις 24 Μαρτίου είναι η επόμενη συνάντησή μας. Αυτή η συνεδρίαση έφτασε στο τέλος. Σας ευχαριστώ.